όσον αφορά την πράσινη βίβλο που σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο παρακολουθείται με τα μεγάλης προσοχής σε πολλές χώρες και σε διάφορους τομείς και στη χώρα μου βεβαίως παρακολουθείται με ενδιαφέρον. Θα δώσουμε το λόγο καταρχάς στην κυρία Πατράο Νέβες για ένα τετράλεπτο που είναι η συγγήτρια. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω και 50 αλληλείς, μια ομάδα που θα μπαίνουν όπου να ναι θα μπουν, πρέπει να μπαίνουν στο ημικύκλιο τώρα, για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής Αλληλείας που εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά πάνω σε αυτή την έκθεση και θέλω να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο και που συζητείται η έκθεση στην Ολομέλεια και παρουσιάζεται στην Ολομέλεια σήμερα. Η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι εμβληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεννήθηκε με μεγάλη δυσκολία Γεννηθήκε τη δεκαετία του 80, πέρασε την πρώτη μεταρρύθμισή της το 2002 και όπως όλοι γνωρίζετε κάποια από τα βασικά προβλήματα όσον αφορά την αλληλεία και το αλληλευτικό δυναμικό, τη γύρανση των στόλων, όλα αυτά τα αρχικά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, να υφίστανται σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί εκ νέου η κοινή αληφτική πολιτική και θα πρέπει η μεταρρύθμιση να είναι ευρεία και εις βάθος. Το περιμένει αυτό ο αληφτικός τομέας επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσει ο τομέας το περιγράφουμε αυτό στην έκθεση. Λέμε ότι πρέπει να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ αλληλεία και περιβάλλοντο και μεταξύ και των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών πτυχών. Σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να εγγυηθούμε την ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων κοινωνικά να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση του επαγγέλματος και οικονομικά θα πρέπει να συνεχιστεί η ύπαρξη του τομέα επιβιωσίμου οικονομικής βάσης. Χωρίς να πετύχουμε αυτούς τους τρεις στόχους ε, ο τομέας δεν θα είναι βιώσιμος εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές αρχές. Ταυτόχρονα θέλουμε οι αλληλείς να ψαρεύουν λιγότερο, να κερδίζουν περισσότερο και να διατηρήσουν τα Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Κάποιε στοιχείε βασικέ αναφέρονται στην έκθεση. Αναφέρουμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε αποκέντρωση του τομέα, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δύναμη που έχουν οι αλλοί οι ίδιοι για την εφαρμογή τη αλληλευτική πολιτική και για τη λήψη αποφάσεων, να λαμβάνουν τι δικέ του αποφάσει πιο κοντά στο, στους ντόπιου πληθυσμούς πρέπει και θα πρέπει οι αποφάσει να λαμβάνονται πιο κοντά στι παραλίε και όχι σε κεντρικό επίπεδο. Να μπορούν να χειρίζονται την πολιτική καλύτερα οι αλληλεί. Θα πρέπει να διοργανώσουν του εθνικού στόλου και του βιομηχανικού στόλου βάσει των προαναφερθισών αρχών και θα πρέπει να έχουμε μοντέλα διαχείριση που να προσαρμόζονται καλύτερα στις διάφορε περιοχέ αλίες και στα διάφορα είδη αλίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και τι αγορέ για τα προϊόντα τη αλίας θα πρέπει να συγκεντρωθούμε επί των αλληλευτικών προϊόντων που έχουν προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να πετύχουμε καλύτερε τιμέ για του αλληλεί όταν πουλάνε τα ψάρια του, θα πρέπει να έχουμε και έναν κατάλογο των βελτίστων πρακτικών και θα πρέπει να εγγυηθούμε, να εγγυόμεθα ε, πολύ υψηλά επίπεδα υγιεινής για όλους τους τόλους, ούτως ώστε να έχουμε γενικά έναν τομέα βιώσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βιώσιμο τομέα αλληλευτικό. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες της μεταπητικής βιομηχανίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των γυναικών στον τομέα τον αλλιευτικών. έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η εισαγωγή αλλιευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πιστοποιείται και υπόκειται στις ίδιες συνθήκες όπως και τα κοινοτικά αλλιεύματα. Μέγεθος αλλιευμάτων, μέγεθο ψαριών που γίνονται δεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Για να χρησιμοποιήσουμε πλήρω το δικό μα δυναμικό πριν εισάγουμε ε, αλλιεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδη, αυτή η έκθεση είναι προϊόν κοινών προσπαθειών όλων των συναδέλφων τη Επιτροπή Αλληλεία ιδίως των σκιωδών εισηγητών με τους οποίους ε, εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη, τη γραμματεία της Επιτροπής τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλους όσους εργάστηκαν πάνω σε αυτή την έκθεση, κυρίως το δικό μου προσωπικό. Είναι μια ομαδική προσπάθεια αυτή η έκθεση και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να την υιοθετήσει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα. το λόγο έχει ο κύριος Μάρτιν Φραγκέιρο από την Ισπανική Προεδρία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η Προεδρία χαίρεται που γίνεται η συζήτηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αποτελεί μια σημαντική, σημαντική συμβολή στην ευρύτατη διαδικασία διαβούλευση, διαβούλευσης που έχει γίνει για την Πράσινη Βίβλο. Οι θέσεις του Κοινοβουλίου ασφαλώς και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την κατάρτιση των νομοθετικών της προτάσεως και από το Συμβούλιο ασφαλώς. Το Συμβούλιο θα εξετάσει εκτενώς όλες τις τοποθετήσεις του Κοινοβουλίου. Και ανάλογα θα ελεγχθούν, θα εξεταστούν και οι νομοθετικές προτάσεις στα πλαίσια της διαδικασίας της συναπόφασης. Κατά το 2009 καλύφθηκαν αρκετές ατέλειες ε, Τη κοινή αλληλευτική πολιτικής λήφθησαν πολλές ε, βραχυπρόθεσμες αποφάσεις, αλλά λείπει από τον τομέα ένα συνολικό πλαίσιο. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να αντιμετωπιστούν αυτέ οι διαρθρωτικές ε, ελλείψεις. Και μιλάμε για πραγματικά ζητήματα όπως διαφοροποιημένοι κανόνες για τους στόλους, οι ποσοστώσεις οι απορρίψεις, η ενσωμάτωση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής στο γενικότερο πλαίσιο της ε, θαλάσσιας πολιτικής, η δημοσιονομική διάσταση και φυσικά και εξωτερική διάσταση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Στα μεμονωμένα κράτη-μέλη, όπως και στο Συμβούλιο συνολικά, εξετάζονται όλες οι πτυχές των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε το 2009. Η Κομισιόν έλαβε 170 προτάσεις και διεξήγε 125 συναντήσεις και από το Σεπτέμβριο του 2010 οι συζητήσεις θα εστιαστούν πλέον στην σύνοψη των διάφορων ιδέων που θα προταθούν. Σήμερα λαμβάνει η χώρα ένα σεμινάριο για την ε, ε, μικρού χαμηλού επίπεδου αλληλεία και για το αλληλευτικό ταμείο, το Ευρωπαϊκό Αλληλευτικό Ταμείο, το οποίο θα καλυφθεί από τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές στις 2-3 Μαΐου θα διοργανωθεί από την Ισπανική, στην, από την Ισπανική Προεδρία συνέδριο στην Λακορούνια αναφορικά με την χρηματοδότηση της αλίας. για τα μικρά και μεγάλα ψάρια. Και στο Βίγκο θα ακολουθήσει εξέταση του σχετικού εγγράφου εργασίας. Η τρίτη φάση, όπως ανέφερα, η οποία θα λάβει χώρα στο δεύτερο ημισή του 2010 θα είναι μια λευκή βίβλος και τέσσερις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται και τα χρηματοδοτικά μέσα. Η αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2013. Το Συμβούλιο βάσει των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το έτος 2011 θα υποβάλει δεσμευτικέ ε, νομοθετικέ προτάσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα. Να ακούσουμε την Επίτροπο, την οποία και καλωσορίζουμε ε, θερμά εδώ στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά ε, η οποία βρίσκεται εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο, την κυρία Δαμανάκη. Εγώ σε κάθε περίπτωση πρώτη φορά είμαι πρόεδρος συζήτηση, σε συζήτηση στην οποία παρευρίσκεται. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ. Και χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ σε μια συζήτηση η οποία έχει τόσο μεγάλη σημασία. Παρακαλώ. Good morning, Mr. President. Thank you for your... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Επειδή είναι η πρώτη μου φορά που παίρνω το λόγο ως Επίτροπος προς τα μέλη του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα και ε, για να συζητήσουμε την μεταρρύθμιση της κοινή αλευτικής πολιτικής, το οποίο αποτελεί θέμα σημαντικό για όλο τον κλάδο. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Νέβε, την εισηγήτρια, για τις σκληρές προσπάθειες που κατέβαλε να συγκεράσει διάφορες απόψεις και να τις συνενώσει σε συνεκτικά έγγραφα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι ελλείψει της πολιτικής μας. όπω ξέρετε, η τελευταία μεταρρύθμιση το 2002 δεν ε, ήταν αρκετά επιτυχη. Και τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα χάσματα για να σημειώσουμε καλύτερα επιτεύγματα στον οικονομικό, κοινωνικό τομέα. Η δημόσια διαβούλευση κατέδειξε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη προς την μεταρρύθμιση αυτή. Φυσικά σήμερα δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα τα θέματα τα οποία θίγετε στην έκθεσή σας. Ωστόσο, λαμβάνοντα υπόψη τις ε, συμβιβαστικές αστροπολογίες για την βιωσιμότητα, την υπερπαραγωγή, τα μικρά και μεγάλα ψάρια, την κατάργηση των απορρίψεων, την σταδιακή εισαγωγή νέων συμφωνιών. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επικοδομητική σας συμβολή. Θα ήθελα να τονίσω δύο συγκεκριμένα θέματα. Καταρχάς, ό,τι αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε, να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην στοχοθέτησή μας για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, να μην υποστηρίζουμε απαραίτητα την κατασκευή νέων σκαφών. Να στηρίξουμε καλύτερα ανταυτού την κοινοτομία, προκειμένου να ανταποκριθούμε στι νέε προκλήσει. Συμφωνώ επίση ε, με αυτά που λέτε για την κοινωνική διάσταση. Θέλουμε να υπάρχουν ασφαλείς θέσεις εργασίας, κλικιστικές θέσει εργασία στην Αλία. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να ακούσουμε τι προτάσει σα και να τι λάβουμε υπόψη. Να σα ενημερώσω ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μα. Θα προετοιμάσουμε μια σύνοψη, μια έκθεση σύνοψης για τις διαβουλεύσεις του προηγούμενου έτους που θα μας βοηθήσει να ετοιμάσουμε τις νέες νομοθετικές προτάσεις. Διοργανώνουμε εργαστήρια για να συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα με τους εμπλεκομένου φορείς και με τη βιομηχανία, τον κλάδο. Από την Ισπανική Προεδρία θα γίνει μια ευρεία σύνοδος τον Μάιο. Θα διοργανωθεί μια ευρεία σύνοδος τον Μάιο και ξέρω ότι, όπως αναφέρατε κι εσείς, ε, λαμβάνει η χώρα σήμερα ένα εργαστήριο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη. Και λυπάμαι που δεν μπορείτε να συμμετάσχετε γιατί έχει τριγωνωθεί εδώ και πολύ καιρό και θα προσπαθήσω στο μέλλον να μην υπάρχει τέτοια επικάλυψη ε, εργασιών στο βαθμό του δυνατού ασφαλώς. Και βάσει όλων αυτών των στοιχείων θα ξεκινήσουμε στο 2010 να προετοιμάζουμε την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα είναι έτοιμη την άνοιξη του 2011. Ελπίζω να είναι πάρα πολύ επικοδομητική η συζήτηση μαζί σας και εσείς ως συνομοθέτες στη συνέχεια θα καλυφθείτε να διαδραματίσετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, να διαδραματίσετε τη νέα πολιτική από κοινού με το Συμβούλιο και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να ακούσουμε τους διάφορους ομιλητές εξ ονόματος των διάφορων ομάδων. Έχουν ζητήσει το λόγο παραπάνω από 30 ομιλητές. Πολύ ιδιαίτερο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους ομιλητές να τηρήσουν το χρονικό όριο που τους ε, δίδεται. και όσοι δυστυχώς ε, ε, υπερβαίνουν το χρονικό τους όριο θα πρέπει να τους διακόψουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εξ του ΕΛΚ, ο συνάδελφος Αντινόρο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και να ευχαριστήσω για την Επίτροπο που παίρνει το βάπτισμα το πυρό σήμερα. Θα έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Είναι σημαντικό αυτό που ε, κάνουμε και θέλουμε αυτή η πράσινη βίβλος που αρχίζουμε να συζητάμε σήμερα αργότερα, όμως να μην γίνει αυτό που έγινε το 2002. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε συνθήκες διαφορετικές. Έχουμε τη συναπόφαση, έχουμε τις συνθήκες της αγώνας Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε θετικά όλα αυτά για να πετύχουμε τους στόχους. Τα βασικά σημεία τα περιέγραψε η συγγήτριά μας, η κυρία Νέβες ε, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν ομάδα του ΕΛΚ, την κυρία Πατράου Νέβες για τη δουλειά που έκανε και που συνάθρισε όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά που πρόθεσε και όλα αυτά που κατάφερα συμπυκνώσει. Θα ήθελα απλώς να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να μπω εντός της αλληλείας βγαίνοντας και λίγο πιο πέρα από αυτά που αναφέρεται στην Πράσινη Βιβλίο τον Ιούνιο που θα, τι θα γίνει στη Λευκή Βίβλιο, την ανάγκη που υπάρχει στις θάλασσε τη Ευρώπης, ανάγκες που υπάρχουν κυρίω και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Σήμερα έχουμε την ανάγκη να θεσπίσουμε κανόνες και να δώσουμε κανόνες στους αλληλεί και στην οικονομία μας. Έχουμε δώσει και κανόνες εδώ και χρόνια, αλλά πάρα πολύ συχνά οι, χώρες, οι παραμεθόριες της Ευρώπης δεν σέβονται τους κανόνες και αντιμετωπίζουμε ένα παράδοξο. Δηλαδή στου αλληλεί μα επιβάλλονται όλα αυτά τα μέτρα και άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ρόλο διαφορετικό. Έχει έναν Υπουργό Εξωτερικών, έχει πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε ένα κοινοβούλιο πιο ισχυρό. Η ευχή είναι ότι όλο η Λευκή Βίβλο, πριν φτάσουμε στη Λευκή Βίβλο, αν μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τι άλλε χώρε με τις τρίτες χώρες, εκείνες που δεν ανήκουν στην Ένωση, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιους κανόνες κοινούς, για ώστε σε όποιον επιβάλλονται οι κανόνες να μην αισθάνεται προδομένο, να μην αισθάνεται προδομένο από την Ένωση και να μην βλέπει την Ένωση περισσότερο σαν εχθρό από τη Σαφίλο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφε. Για τρία λεπτά η κυρία Αντρέ έχει, το έχει το λόγο εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, λοιπόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της του Συμβουλίου και την κυρία Δαμανάκη. Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση σε ό,τι αφορά την αλληλεία. Θα πρέπει να ορίσουμε ποιε θα είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ οι οποίε θα εγγυηθούν τη βιωσιμότητα τη αλληλεία. Αλλά παράλληλα, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό προϊόν το οποίο έχει βαρύνουσα σημασία για τις χώρες μας από πολιτισμικής, πολιτιστικής άποψης αλλά και από οικονομικής άποψης. Θα ήθελα να πω προς την κυρία Δαμανάκη ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία προκύπτουν το 2002. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα νέες μορφές ε, οικονομικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, οι οποίες θα ταιριάζουν καλύτερα στο σύστημά μας, γιατί παρουσιάστηκαν προβλήματα με τις ποσοστώσεις και για τις απορρίψεις. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσουν αυτές οι περίφημες ε, απορρίψεις, ούτε για τους αλληλείς, αλλά ούτε για το μέλλον του πλανήτη. Θα πρέπει η μεταρρύθμιση να εγγυηθεί μια βιώσιμη αλληλεία, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι θα επιτρέψει την ευέλικτη προσαρμογή στις διάφορες ε, καταστάσεις που θα προκύψουν και θα πρέπει φυσικά να λεφθούν υπόψη και τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Και η παρακτία αλληλεία, ε, η παρακτή αλληλεία θα πρέπει να διαμορφωθεί φυσικά διαφορετικά από τη η αλληλεία ανοιχτή θάλασσα. και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώς θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν θέματα όπως η παράνομη αλίευση, η εισαγωγή ηχθείων από τρετές χώρες. Χρειάζεται μία εναρμόνιση των κυρώσεων. Χρειαζόμαστε ε, διεθνείς συμφωνίες σε ό,τι αφορά την τήρηση των συμφωνίων και χρειαζόμαστε και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυηθεί καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα από τη φυστάμενη πολιτική. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να λάβουν μια αναγνώριση, μια αναγνώριση του επαγγέλματό του. Και θα πρέπει να έχουν και την οικονομική δυνατότητα να επιβιώσουν. Και ακριβώς αυτό το, αν θέλετε, μη ορατό κομμάτι των άλλων θα πρέπει να βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να σας πω ότι η μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής δεν είναι μόνο ένα νομοθέτημα, είναι ένα σημαντικό τμήμα της μεταρρύθμισης όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας των θαλασσών και όλου του κόσμου. Θα πρέπει φυσικά να επιδείξουμε και θάρρος. Θα πρέπει να ασκήσουμε μια πολιτική χωρίς φόβο, με τόλμη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως έχει και φυσικά θα πρέπει να βρούμε ε, μια ισορροπία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου. Σας ευχαριστώ κύριε Άντρες, εξ των Φιλελευθέρων. Δύο λεπτά, ο κύριος Χάγκλοντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για εκείνους από εμά που εργαστήκαμε σκληρά πάνω σε αυτή την έκθεση, είναι καλό συνέστημα το ότι φτάσαμε μέχρι τον Ολομέλεια. Και εν είδη εισαγωγή θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά την εισηγήτρια για την έξοχη δουλειά που έκανε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η κοινή αληφτική μα πολιτική χρειάζεται μεταρρύθμιση. Όσον αφορά την ομάδα των φιλελευθέρων, θεωρήσαμε σημαντικό να ξεκινήσουμε από μια προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση. Αλλά όπως αντιμετωπίζεται το θέμα από την έκθεση, νομίζω ότι είναι καλή η προσέγγιση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα όπως είναι οι απορρίψει και το υπερβολικό δυναμικό που υπάρχει, αλληλευτικό δυναμικό. Και γι' αυτό χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία για σχετικά μέτρα, διότι Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική για τις απορρίψεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να δικαιολογηθεί. Άλλο θέμα είναι η περιφερειοποίηση της κοινή αληφτικής πολιτικής. Είναι σημαντικό οι αποφάσεις να λαμβάνονται και να εκτελούνται σε περιφερειακό επίπεδο, διότι ποικίλουν οι καταστάσεις ευρέως, ανάλογα με την περιοχή της Ευρώπης που εξετάσεις. Μια άλλη ευπρόσδεκτη μεταρρύθμιση είναι η ιδέα για την εισαγωγή μιας ξεχωριστής προσέγγισης για την παράκτη αλληλεία μικρής κλίμακας. Αυτό είναι κάτι που ενδιέφερε ιδιαίτερα την ομάδα των φιλελευθέρων. Σαν Φιλανδός που ζω κοντά στη Βαλτική, χαίρομαι ιδιαίτερα που οι μεγάλοι πληθυσμοί το, της φώκιας και των κορμοράνων λαμβάνονται υπόψη, διότι ε, απειλούν όλους ιδιαίτερους αυτά τα ζώα την ε, αλία στην περιοχή οι ελευτικέ μετά συμφωνίε με τρίτε χώρε ε, αυτό αφορά και τι πολιτικέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταιριάζουν αυτά τα δύο. Η συμφωνία με τη Γουινέα ε, είναι κάτι καλό, είναι καλό παράδειγμα, διότι την καταψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία και δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Ε, νομίζω ότι έχουμε ένα καλό έγγραφο, είναι μια καλή αφετηρία και νομίζω ότι μπορούμε να βλέπουμε προς το μέλλον σε καλύτερη και βελτιωμένη πολιτική αλίας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους των Πρασίνων για δύο λεπτά, δυόμιση λεπτά, η κυρία Λοβίν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπη, κυρία Δαμανάκη. Όταν άρχισα να εξετάζω στην αρχή την κοινή ελευθερική ε, πολιτική και τις καταστροφικές συνέπειες της το 2002, στη Σουηδία και στο Σουηδικό Κοινοβούλιο τότε μία μειονότητα στο κοινοβούλιο ήθελε να σταματήσει την αλληλεία του βακαλάου. Παρά το γεγονός ότι οι Σουηδοί ψαράδες αποζημιώθηκαν διότι σταμάτησε η αλία του μπακαλιάρου, εάν απαγορευτεί τελείως αυτή η αλία, θα πρέπει να εξεταστούν και οι συνέπειες που έχει αυτή η απαγόρευση της αλίας του βακαλάου ε, στα αποθέματα του βακαλάου στη Σουηδία θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της υπερβολικής αλίας, της υπεραλίας. Θεωρήθηκε ότι συνέβαλε στο πρόβλημα και η Σουηδία λόγω υπεραλίας. Το 2002 έγινε η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής και έπρεπε στα πλαίσια αυτά να αναγνωριστεί ότι τα σκάφη ε, ήταν ε, υπερβολικά αποδοτικά όσον αφορά την αλληλεία. Είχαν υπερβολική απόδοση. Και όσο μιλάμε για τον ερυθρό τόνο που συζητήσαμε και ποια είναι η κατάσταση στη Μεσόγειο όσον αφορά τον ερυθρό τόνο από το 2005 και μετά εξετάσαμε αυτό το θέμα και 34 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για να βελτιωθούν οι αληφτικοί στόλοι η αποδοτικότητα των στόλων. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και πρόβλημα υπεραλίευσης. Λοιπόν, και 5,4 εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για τον αφοπλισμό, αν θέλετε, για τον παροπλισμό σκαφών. Θα πρέπει να γίνει μια ριζική μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής. Θα πρέπει το όλο θέμα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από τα σκάφη να εξεταστεί και αυτό το θέμα. Πρέπει να προσέξουμε τα αποθέματα των ε, ψαριών που είναι πολύ σημαντικά για όλους τους ψαράδες και κυρίως και για τους ψαράδες Αφρικής. Υπάρχει μια παράγραφος που δεν μου αρέσει σε όλη την έκθεση. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι καλά. Εκεί αναφέρεται στην εξωτερική αλληλευτική πολιτική που προστατεύει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Αλίας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το υποστηρίζουμε σαν πολιτική του 2010. Ευχαριστώ κυρία Λαβίν. Και τώρα εκ μέρου τη ομάδα του, τη ECR, για δύο λεπτά, ο κύριο Γκρομπάρτσικ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την κυρία, την προηγούμενη ομιλήτρια, για την ε, συμβολή της. Χρειαζόμαστε μεγάλη αποφασιστικότητα εδώ και μεγάλη, ε, μεγάλο θάρρος για να καταρτήσουμε μια τόσο καλή έκθεση. Αυτή η έκθεση αποτελεί μια βάση για την οικοδόμηση της μελλοντικής αλευτικής πολιτικής, η οποία χρήζει βαθιάς μεταρρύθμισης για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες, ε, στα μελήματα των περιβαλλοντικών διαστάσεων αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πρέπει στη διαδικασία αυτή να έχουμε απελευθέρωση της αγοράς και θα πρέπει να ισχύσουν οι όροι που είναι απαραίτητοι. Λαμβάνοντας ε, υπόψη τις απόψεις τις επιστημονικές αλλά και του κλάδου. Η νέα αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να δώσει μια νέα όθηση για την ανάπτυξη της πολιτικής αυτής σε μια Ευρώπη η οποία πλήττεται από την κρίση. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υγιή ψάρια για τα ηχθιάλευρα και να απομακρυνθούν τα τοξικά αλλιεύματα από το τραπέζι του Ευρωπαίου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε ιδιαίτερα και χρειάζεται ένα δίκαιο σύστημα για την αλλιεύση το οποίο θα αντικαταστήσει το σύστημα των ποσοστώσεων, το οποίο επιδέχεται καταχρήσεων. Και αυτό για όλες τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση αυτή και ελπίζουμε να τροποποιηθεί το σύστημα το υφιστάμενο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εξ ονόματος της ομάδας της ΓΚΟΕ, δύο λεπτά, η κυρία Φρέιρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, στην πράσινη βίβλο σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να είναι δημιουργική, προσπαθεί να εφεύρει ένα σύστημα μεταφοράς αλληλευτικών δικαιωμάτων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ιδιωτικά δικαιώματα αλίας. Αυτή η πρόταση απερίφθη στην πρώτερη μεταρρύση. Δέκα χρόνια αργότερα επανέρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την πρόταση για την πώληση αλληλευτικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια ιδιωτικοποίηση των αλληλευτικών πόρων ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι ισχυροί φορεί, ισχυρέ επιχειρήσει θα μπορούν να ασκήσουν αυτή την εξουσία του αγοράζοντα αλληλευτικά δικαιώματα σε περιοχέ που ε, στην οποία ασχολούνται οι αλληλείς μικρής κλίμακας και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημα αποτελέσματα στις ακτές ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα είναι πρόβλημα για τους ντόπιου ψαράδες. Είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πρόταση. Αυτή η πρόταση επουδενή δεν εγγυάται τη βιωσιμότητα των αλληλευτικών αποθεμάτων. Εάν πωλήσουμε δικαιώματα σε περιορισμένο αριθμό εταιριών, αυτό δεν σημαίνει ότι η αλληλευτική προσπάθεια θα μειωθεί, απλώς ότι η προσπάθεια αυτή θα συγκεντρώνεται υπερβολικά σε κάποιες περιοχές όπου έχουν πωληθεί τα δικαιώματα. Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε δικαιοσύνη σε αυτόν τον τομέα. Αυτό σημαίνει παρέμβαση στην αγορά, καλύτερα συστήματα αγοράς για, για τον τομέα και καλύτερες τιμές για τα ψάρια. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε δίκαιη κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε όλη την παραγωγική αλυσίδα από τον αλία μέχρι το εργοστάσιο μεταπητική βιομηχανία μέχρι το μαγαζί. Είναι σημαντικό λοιπόν η διαχείριση των αλλιευτικών αποθεμάτων γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Είναι αντίθετο προς το κεντρικό σύστημα το πλαίσιο που δημιουργείται δηλαδή από τη συνθήκη της Λισαβόνας που δίνει αποκλειστικά δικαιώματα διαχείριση των λευτικών αποθεμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, κάθε παραλίας, κάθε στόλου, κάθε κοινότητα να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την εξέβρεση λύσεων για τον αληφτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι πολύ διαφορετικό αυτό το σύστημα από, μια, από ένα κεντρικό σύστημα. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριο Μπάφτον που θα μιλήσει εκ μέρου τη ομάδα του. Την Ευρώπη τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην κυρία ε, Δαμανάκη να, το άρθρο, για το άρθρο 47 η την κοινή αλληλευτική πολιτική να λάβει υπόψη τη Βρετανία. Διότι και επίση και το ψάρεμα με το αγκίστρι, το ε, τεχνικό συμπεριλαμβάνεται, με το καλάμι. Ε, θα υποτίθεται θέλουμε να προστατεύσουμε τα ληφτικά αποθέματα. Ήταν ανεπιτυχή η κοινή ληφτική πολιτική για τη βιωσιμότητα. 91% των ληφτικών ε, αποθεμάτων ε, θα έχουν υπεραληφθεί μέχρι το 2015. Δεν είναι... Τι... πώς γίνεται, ας πούμε, άμα με μεγάλες στράτες που αλλιεύουν όλα τα ψάρια είναι κακό. Και το αντίθετο τη βιωσιμότητα είναι να ψαρεύει κανεί ψάρια, να μην τα αρέσει και να τα πετάει ξανά στη θάλασσα. Όμω με το παραγάδι όταν ψαρεύει κανείς τεχνικά, δεν βλάπτεται. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι ε, ψαρεύουν έτσι στο Βρετανία και περίπου 2, δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο τζίρος. 13.000 ε, επιχειρήσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία ασχολούνται με τον τομέα αυτό του ψαρέματος ως τεχνικού. Λοιπόν, αυτοί οι ψαράδες παίρνουν και ψαρεύουν μόνο αυτά που θέλουν να φάνε και αφήνουν τα μικρά νέα ψάρια να μεγαλώσουν και ρίχνουν πίσω εκείνα που δεν χρειάζονται τα ψάρια. Σε κάποιες περιπτώσεις έτσι, με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στα προγράμματα συντήρηση. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτό που θέλει, θα υποχρεώνονται να εκφορτώνουν ό,τι πιάνουν και να μετράει ποσόστοσή του και να συγκρίνεται με την εθνική. Λοιπόν, αυτό το ψάρεμα το είναι οικολογικά σωστό και αν ασχολούνται με αυτό περισσότεροι άνθρωποι, θα μειωθεί η ε, ζήτηση για το εμπορικό ψάρευμα που απειλεί πολλά είδη. Η κοινή ελευτική πολιτική πάντα ε, ήταν εναντίον του Βρετανικού στόλου που επιτρέπεται να ψαρεύει μόνο το 7% του βακαλάου και ένα πέμπτο της ποσόστοσης στα δικά μα χωρικά ύδατα. Ίσως η Επίτροπος θα ήθελε να υποστηρίξει τους ερασιτέχνες αλληλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον ίδιο τρόπο όπως ο προκάτοχός τη έδειξε ευαισθησία στις ανάγκες των αλληλείων της δικής του χώρου όταν επέβαλε την αγόρευση της αλληλείας του ερυθρού τόνου που ήταν 200 εκατομμύρια ο τζίρο ευρώ το χρόνο για τη Μάλτα. Λοιπόν, θα είπα να προσέξουμε του πόρου. Οι ερασιτέχνου ψαράδε ψαρεύουν το 1% των αλλιευμάτων που απομένουν μόλι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διστάζει να προστατεύσει ήδη που κινδυνεύουν, αλλά θέλει να ρυθμίσει και το ψάρεμα τη αναψυχή. Οπότε θα πρέπει αυτό να το προσέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Τελειώνουμε αυτό τον γύρο των ομιλητών εκ μέρου των ομάδων του και δίνουμε το λόγο στην κυρία Ντότ που θα μιλήσει για 1,5 λεπτό εν ονόματι των μη εγγεγραμμένων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην ε, Βόρεια Ιρλανδία και στη σχετική αλληλευτικό κλάδο 27 χρόνια αλλαυτικής πολιτικής τελικά κατέληξαν στην παράγραφο 138 της έκθεσης αυτής που επαναλαμβάνει ότι λίγους από του τομεί ε, όπου σημείωσε επιτυχία η κοινή πολιτική είναι όπου τα κράτη-μέλη διατήρησαν τον έλεγχο. Το ιδανικό για μας θα ήταν να διαγραφεί η κοινή ελληνική πολιτική ή να αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από αυτή. Και έτσι τα κράτη-μέλη να έχουν και πάλι τον έλεγχο των υδάτων του. Δυστυχώ δεν ζούμε σε αυτόν τον ιδανικό κόσμο. Η μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική αναμφίβολα θα καταλήξει σε μια λύση η οποία δεν θα είναι η καλύτερη για του αλληλείς τη Βόρειας Ιρλανδία. Μια λύση η οποία όπω και τα τελευταία χρόνια θα χαρακτηρίζεται από την παρακμή τη ελευτικής δραστηριότητα και των αλληλευτικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται ο κλάδος μας το οποίο κατέδειξε και η Πανολευθρία ε, του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Δεν θα είναι λοιπόν η καλύτερη λύση αυτή, αλλά υποστηρίζω την περιφερειακή διάσταση και την περιφερειακή διαμόρφωση της κοινής πολιτικής και υποστηρίζω ότι θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις αρχές ε, η κοινή πολιτική στις διαθάσεις, στις οικονομικές, τις και τις οικονομικές. Θεωρώ ότι μια πολιτική η οποία θα ανατρέψει τις ε, καταστροφικές συνέπειες της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Ωστόσο θεωρώ ότι κάποιες από αυτές τις ριζοσπαστικές αλλαγές οι οποίες υπόσχεται, τις οποίες υπόσχεται η έκθεση θα καταλήξουν σε εκ νέου παρακμή του στόλου. Ευχαριστώ κυρία Ντός. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές που μιλούν ε, για λογαριασμό τους να τηρείτε το χρονικό σας όριο, παρακαλώ. Καταρχάς, λοιπόν, δύο λεπτά η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρα, στη μεταρρύθμιση αυτή. Δεν καταφέραμε και δεν έχουμε πετύχει όλα όσα θέλαμε. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε και να διαμορφώσουμε εκ νέου την πολιτική αυτή. Ιδάλλως θα είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι για την πανελευθερία Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, λοιπόν. Και συχνά ασκείται κριτική στο Κοινοβούλιο για το σύστημα αυτό που απέτυχε, για την διατήρηση των αποθεμάτων και για την ισορροπία στον κλάδο. Δεν είναι λοιπόν εύλογο να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, γιατί ήδη έχει συζητηθεί στο Κοινοβούλιο το θέματα των ποσοστώσεων και τα αποτελέσματα των προσπάθειών ε, του αλευτικού κλάδου. Στην έκθεση αναφέρεται ότι ότι δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές και διάφορες λύσεις. Αυτό ωστόσο περιέχει και μία αντίφαση, την οποία δεν κατανοώ. Γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί και να αξιοποιηθεί ένα μέσο το οποίο θα προδιαγράφει τα ίδια για όλους. Γιατί μιλάμε για τους αλληλείς, δεν μιλάμε μόνο για μια διαρκή επιδότηση. Η αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να εγγυάται τον ανταγωνισμό και σίγουρα θα πρέπει να επιτρέπει την ε, καλή λειτουργία των αγορών. Χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική. Δεν μπορούμε η εμπορική πολιτική και οι κανόνες προέλευσης στις νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και η ανταγωνιστικότητα να καταστρέψουν την ανταγωνιστικότητα του αλευτικού κλάδου και θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα των τρίτων χωρών. Νομίζω ότι όλα αυτά επιβαρύνουν τον αλευτικό μας κλάδο. Είναι καλή η συνένεση, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε πέρα από αυτή, γιατί σίγουρα θα παραμείνουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα καλύθουμε να επιλύσουμε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δύο λεπτά κυρία Ροντέστ. Ευχαριστώ συνάδελφοι Αξιότιμη κυρία Επίτροπε Δαμανάκη, σας καλωσορίζουμε και καλωσορίζουμε και όλους τους αλληλείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια ημερομηνία ορόσημο. Μετά την ε, επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας, για πρώτη φορά τοποθετούμαστε για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Έχουμε πολύ ευθύνη να αναλάβουμε τις επόμενα, τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ καλή η έκθεση και ευχαριστώ και την κυρία εισηγήτρια για την έκθεση της. Είναι σημαντικό να περάσουν οι δημοκρατικές αρχές στην έκθεση και σε αυτές συγκαταλέγεται και η υποστήριξη των, της αλληλευτικής δραστηριότητας. Οι μικρές ε, αλληλευτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη υποστήριξη και θα πρέπει στις παράκτιες περιοχές ε, όχι μόνο να τονιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά και η τουριστική δραστηριότητα. Θα πρέπει να βελτιωθούν κάποια τμήματα της ε, νομοθεσίας και έχουμε υποβάλει σχετικές προτάσεις. Θέλουν να διευκρινίσουν οι σοσιαλδημοκράτες ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η υπεραλίευση. Και αυτό α, επηρεάζει και την οικολογική βιωσιμότητα, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα. Άρα η οικολογία θα πρέπει να λάβει προτεραιότητα. Τρίτο βασικό σημείο είναι η εξωτερική δραστηριότητα, της, η εξωτερική διάσταση συγγνώμη, της κοινής αλληλευτικής ε, πολιτικής. Θέλουμε να διαγραφεί η παράγραφος 121 αναφορικά με τα τρίτα κράτη. Θα πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στα ευρωπαϊκά ύδατα όπως και στα δικά του ύδατα, στα δικά του χωρικά ύδατα. Να προωθήσουμε λοιπόν την δημοκρατία και την αγορά και να φροντίσουμε να μην ε, ε, καταδικαστούμε από ε, δικτατορίες διεφθαρμένες. Και τέλος, να πω το εξή ότι υπάρχουν πάρα πολλά εθνικά συμφέροντα που είναι αντικρουόμενα στην κοινή πολιτική και αυτό φυσικά δεν αποτελεί μυστικό και οδήγησε σε έντονε συζητήσει μεταξύ των ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταφέραμε να βρούμε έναν καλό συμβιβασμό. Όταν θα προκύψει λοιπόν η νομοθεσία θα πρέπει να εστιαστούμε ακόμα πιο έντονα στην εξέβρεση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων και να αφήσουμε στο Συμβούλιο τις, μικρο, τις μικρές ε, εθνικές ε, συμφέροντα. Ευχαριστώ Σκάλαχερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, κυρία Επίτροπε, καταρχάς καλωσορίζω την κυρία Επίτροπο στο Κοινοβούλιο, στην πρώτη επίσκεψή τη στο Κοινοβούλιο, στην πρώτη ομιλία τη και ευχόμαι καλή τύχη στη θητεία τη. Συγχαίρω, και την κυρία Νέβε, τη συνάδελφο, για την ετοιμασία αυτή τη εκθέσεω. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι χρειαζόμαστε καλύτερους στόχους, σαφέστερους στόχους στη νέα κοινή ελευτική πολιτική και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη Οικολογικέ και κοινωνικές αρχές και πτυχές. Χρειάζεται ριζοσπαστική αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετάσχουν και χρειαζόμαστε μια βιώσιμη διαχείριση των αλληλευτικών μας πόρων και ταυτόχρονα είναι ουσιαστικό να υπάρξει βιώσιμη εργασία που θα εξασφαλίζεται για τους αλληλείς της Ευρώπης. Λοιπόν, ε, για τους ψαράδες που είναι στις μικρές ε, παράκτης κοινωνίας μας τεφέρει. για, τις, για την αλία μικρής κλίμακας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η αλία για τις υπερπεριφερειακές περιοχές που δεν έχουν εναλλακτική εργασία. Και ενεθαρρύνθηκα όταν άκουσα την Επίτροπο σήμερα το πρωί που αναφέρθηκε σε αυτό το είδος αλίας. Τα περισσότερα σκάφη που αλλιεύουν σε αυτέ τι περιοχέ είναι μικρότερα από το 15 μέτρα αλλιεύουν ψάρια σε ποσότητες που δεν έχουν μεγάλη συνέπεια και αντίκτυπο όσον αφορά τα αλλιευτικά αποθέματα και βεβαίως πολλοί από αυτούς ε, αλλιεύουν ήδη που δεν είναι στις ποσοστώσεις και πιο σημαντικό δεν έχουν άλλη πηγή εργασίας πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό υπέβαλα μια τροπολογία που ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναγνωρίσει συγκεκριμένα αυτές τις απομακρυσμένες κοινωνίες η εισαγωγή των ΡΑΞ ήταν κάτι επιτυχές, οπότε η σωστή διαχείριση, οι σωστές δομές θα πρέπει να δημιουργήσουν θετικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη υπευθυνότητα από πλευρά των εμπλεκομένων φορέων και, και η δημιουργία μιας κοινής αλευτικής πολιτικής έτσι θα είναι πιο ευαίσθητη και θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες. Η... Μετά το δημοψήφισμα στη χώρα μου εγκρίθηκε, επικυρώθηκε οι συνθήκε τη Αβώνα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα έχει μεγαλύτερε νομοθετικέ ευθύνε. Και ξανά αναγνωρίζει αυτό το γεγονό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπουμε συνεργασία μαζί με την Επίτροπο. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι βασικέ διατάξει τη εκθέσεω θα θα αναφέρονται στι σημαντικέ ε, μεταρρυθμίσει που χρειάζεται στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο ο συνάδελφο Χάουτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπε ο συγητής όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική ότι τα αρχικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται. Συμφωνώ και από 27 χρόνια εμπειρίας που έχω στη Σκοτία όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική είδα ότι η εμπειρία αυτή ήταν κακή εμπειρία. Αν θέλουμε να πάμε σε ένα σύστημα διαχειρίσεως των αλληλευμάτων που λειτουργεί και νομίζω ότι αυτό θέλουμε όλοι να κάνουμε, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να στερνιστούμε μια αντελώς διαφορετική προσέγγιση. Η κεντρική άκαμπτη κοινή ελευτική πολιτική απέτυχε παταγωδό και θα πρέπει να το δεχτούμε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Αντιστρόφω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι τοπική διαχείριση εντό τη ζώνη των 12 μιλίων μέχρι τώρα, μέχρι τώρα υπήρξε επιτυχή. Και αυτό είναι ένα μάθημα. Υπέβαλα τροπολογίε μέσω των οποίων επιδιώκω υποστήριξη από πλευρά συναδέλφων και ζητώ μέσω των τροπολογιών αυτών πραγματικέ εξουσίε να εκχωρηθούν στα κράτη τα αλλιευτικά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών αυτών και των, και των εμπορικών φορέων με τέτοιο τρόπο ώστε ε, να εφαρμόζονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο διάφορα μέτρα βιώσιμη αλληλεία. Και θα πρέπει να διατηρηθούν τα ιστορικά δικαιώματα ε, βάσει τη αρχή τη σχετική σταθερότητα. Πιστεύω ότι αυτοί που έχουν περισσότερα να κερδίσουν από μια επιτυχή διατήρηση των λευτικών αποθεμάτων είναι οι ελευτικέ κοινότητε και τα ελευτικά κράτη και όλοι αυτοί είναι σε καλύτερη θέση να πάρουν τις αποφάσεις περί της διαχειρήσεως και των σχετικών σχεδίων και της εφαρμογής των σχεδίων για τα αλλιεύματα ε, συνεργαζόμενοι σε περιφερειακό επίπεδο. Λοιπόν, είναι θέμα αλληλευτικών αποθεμάτων και των αλλιέων. Δημιούργησε προβλήματα σε αυτά η κοινή αλληλευτική πολιτική και η κοινή γνώμη ε, έχει χειρότερη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη αποτυχία τη ευρω... αλληλευτική πολιτική. Και αυτό διακινδυνεύουμε. Αν δεν πετύχει αυτή η μεταρρύθμιση, κινδυνεύουμε αυτή η εικόνα να αμαυρωθεί περαιτέρω. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κ. Στίβενσον, ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Πατράου Νέβες, την εισηγήτρια για την σκληρή δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή. Έχουμε εδώ μια ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά, να αλλάξουμε κατεύθυνση σε μια πολιτική επί της όλοι συμφωνούν ότι έχει στεφθεί με αποτυχία. Αλλά για να γίνει αυτή η ριζοσπαστική αλλαγή δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντο. Η να σταματήσει η μικροδιαχείριση, να σταματήσει η διακυβέρνηση από πάνω προς τα κάτω και να σταματήσουν οι τιματζίδικες λύσεις. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέλος της πανολευθρίας του κλάδου. Θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα εναρμονιστούν ε, οι παραγωγή του στόλου με τα αποθέματα και θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην αλληλεία AIU και θα πρέπει να δοθεί νέα ουσία στις βασικές αρχές της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, η διατήρηση των αποθεμάτων, η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Μόνο έτσι θα σημειώσουμε πραγματική πρόοδο. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό τώρα στην κυρία Ρόσμπακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής και είναι πραγματικά ε, η στιγμή να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Αλλά θα ήθελα να πούμε το εξή. Τα εχθιαποθέματα στις θάλασσές μας απειλούνται και συμφωνώ απόλυτα με τους πράσινους σε ό,τι αφορά την οικολογική διάσταση. Θεωρώ όμως ότι οι τροπολογίες τους στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητες πραγματικά για να εγγυηθούμε τα εχθιοποθέματα και στο μέλλον τα μέτρα έχουν πραγματική σημασία για το μέλλον. Το θέμα είναι πώς θα διατηρηθεί μια απαγόρευση για την αλίευση των ηχθείων και των οστρακοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια παραγωγής τους. Γιατί όταν ένας βακαλάος ε, όταν ε, γίνεται αλίευση ενό βακαλάου με αυγά, ουσιαστικά τι κάνουμε. Καταστρέφουμε όλη την επόμενη γενιά. Χαίρομαι λοιπόν που το πράσινο βιβλίο αυτό ε, εξετάζει και θέματα παράκτης ε, αλίευσης, γιατί και εκεί θα τεθεί θέμα θέσεων εργασίας. Η πράσινη βίβλος αυτή τονίζει και την βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου όντως να προστατεύσουμε τα ψάρια εκείνα τα οποία ζουν στα ύδατα τρίτων χωρών. Και επίσης έτσι θα προστατευτούν και τα τρίτα. Ο κύριος Μπρόνς, ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ. Το δικό μας το κόμμα πιστεύει ότι η προστασία των αποθεμάτων νυχθείων είναι θέμα κάθε χώρας μέλους. Διότι ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση στα χωρικά ύδατα της χώρας του. Το πρόβλημα βέβαια είναι παγκόσμιο όταν μιλάμε για τα αποθέματα. Όμως αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας με τέτοιο τρόπο ώστε να φροντίσουμε να μην ε, ψαρεύουμε τα μικρά ψάρια στις θάλασσές μας. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια έχουμε φεύρει κάποιος δηλαδή ένα σύστημα με το οποίο τα ψάρια καταφέρνουν τα πιο μικρά να φύγουν και τα πιο μεγάλα για να μην ξεπεράσουμε τις ποσοστώσεις να μπορούν να φεύγουν. Η Επιτροπή είναι κάτι που πρέπει να το λάβει υπόψη της και ολόκληρος ο κόσμος. Δύο λεπτά τώρα, ο κύριος Κάντεκ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Αντίθετα με άλλου, εγώ πιστεύω ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Πράσινη Βίβλο συνεισφέρει σημαντικά και είναι ζωτική σημασία για την εκπόνηση τη νέας κοινή ελευτικής πολιτικής. Είναι μια πλήρης έκθεση η οποία ασχολείται με όλες τις πτυχές, την προστασία των πόρων πρώτα απ' όλα, την ε, κληρονομιά που έχουμε σε αυτό το τομέα και μιλάει για ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Σήμερα εκφράζω την ικανοποίηση της Γαλλίας για την απόφαση αυτή για την πρόταση μάλλον αυτή του Κοινοβουλίου και ευχαριστώ και την Μαρία που βοήθησε πολύ σε αυτή τη δουλειά. Η έκθεση αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη που υπάρχει να ενισχύσουμε την επιστημονική γνώση που διαθέτουμε, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι αποφάσεις αδιαφυσβήτητες. Ναι, πρέπει να προστατεύσουμε τους πόρους, να έχουμε μια βιώσιμη αλεία, αλλά να μην τα βάλουμε με έναν επαγγελματικό τομέα, ο οποίος έχει περάσει πολλά τον τελευταίο καιρό. Ναι, εξελισσόμαστε σε μια οικονομία αγοράς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την οργανωμένη ρύθμιση του τομέα. Χαίρομαι πολύ για τους συμβιβασμούς στους οποίους καταλήξαμε στην Επιτροπή. Πράγματι, δεν αναφέρεται ρητά το, η μετάβαση του δικαιώματος. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης θεωρείται από σαν ε, μια απάντηση σε οικολογικούς, οικονομικούς ε, και, άλλους, και άλλες ανησυχίες του τομέα. Όχι όμως, μια ευρωπαϊκή αγορά χωρίς ρύθμιση δεν είναι κάτι το επιθυμητό σήμερα, διότι θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία. Ακόμα κι αν πρέπει να έχουμε νέα συστήματα διαχείρισης για τη βιομηχανική αλία και εδώ συμφωνώ με την αδελφο, Κάρμεν Φράγα, Παρ' όλα αυτά είμαι πεπισμένο ότι αν διευρύνουμε την διάταξη αυτή και την εφαρμόσουμε πολύ, αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό για τη μικρή κλίμακα αλεία την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε. Κυρία Δαμανάκη, βασιζόμαστε σε εσά για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ένα λεπτό, κύριο Αρσένη τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Επίτροπε Δαμανάκη, κύριε Φραγέρο. Η σημερινή κοινή αλληλευτική πολιτική έχει αποτύχει. Τα περισσότερα αποθέματα καταραίουν. 88 των αλληλευτικών αποθεμάτων αλλιεύονται πέρα από το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο. Το 30 των αλληλευτικών αποθεμάτων βρίσκονται εκτό ασφαλών βιολογικών ορίων, που σημαίνει ότι έχουν πολύ χαμηλέ πιθανότητε να αποκατασταθούν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα, που αλλιεύονται ακόμα και σε ηλικίε πριν την ε, ξεκινήσει η αναπαραγωγική διαδικασία. Η συζητούμενη λοιπόν αναθεώρηση είναι εντελώ απαραίτητη. Η προστασία των αλλιευμάτων είναι προπόθεση για την προστασία των αλλιέων για να αποτρέψουμε την κατάρρευση τη ευρωπαϊκή αλίας είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε την αλληλευτική προσπάθεια και τον ευρωπαϊκό αλληλευτικό στόλο. η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να αποτελέσει την πρωτεύουσα αρχή τη νέα μα κοινή αλληλευτική πολιτική και να συνοδευτεί με το μακροχρόνιο σχεδιασμό συμμετοχικέ διαδικασίε και την εφαρμογή τη αρχή τη πρόληψη. αυτή η μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη διατήρηση των ειδών θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε όλε μα τι διεθνεί αλληλευτικέ συμφωνίε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ να αποφασίσουμε αυτές τις αρχές, τις βασικές αρχές, προκειμένου να αναδειχθεί ένα αποκεντρωμένο και συμμετοχικό σύστημα που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο με τη συμμετοχή των αλλιέων και το σεβασμό στι ανάγκε των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ευχαριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε. Ένα λεπτό τώρα. Η κυρία Ρέιμερς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα βήμα μόνο στο μακρύ δρόμο της μεταρρύθμισης κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους συντονιστές για την έκθεση και για την αποδοτική εργασία. Μιλώ και τάσομαι υπέρ τη εκβάθρων μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτικής, αλλά δεν υπάρχει θάρρο, Είναι πιο σημαντικό να διατηρηθεί η αρχή τη σχετική σταθερότητα. Πέραν τούτου, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους κορμοράνους και να υποδείξω το θέμα της, ε, του σχεδίου διαχείρισης που έχει ήδη ε, τονίσει το Κοινοβούλιο. Η αλληλεία μας έχει οικονομική αλλά και πολιτιστική διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν στην μεταρρύθμιση αυτή της κοινή αλευτικής πολιτικής θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη, να υπάρχει ισορροπία μεταξύ οικονομικών και άλλων διαστάσεων. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό τώρα ο κύριος Βαντάλλον. Μικρό, Πρόεδρε, η βιωσιμότητα δικαίως αναφέρεται ως σημείο κλειδί στην έκθεση. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό για το μέλλον της ε, αλληλείας και για την εγγύηση του, της εξασφάλισης του περιβάλλοντος. Ε, η στοχοθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι καινούργια, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε στους στόχους αυτούς και αυτό τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για μεταρρύθμιση. Και υποστηρίζω την ε, περιφερειακή διάσταση που θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να δώσουμε πιο πολύ περιθώριο στον ίδιο τον κλάδο και να λάβουμε υπόψη και την οικολογία. Γιατί στο παρελθόν είχαμε μια πολιτική η οποία είχε πάρα πολλέ λεπτομέρειες και ήταν αναποτελεσματική. Επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε την καλύτερη τήρηση των ε, κανόνων. Γιατί όποιοι τηρούσαν του κανόνε τελικά ζημιώνονταν. Και είμαι ε, περήφανος για του Ολλανδού αλληλεί, γιατί μαζί με του Δανού είχαν σωστές ποσοστώσεις. Θα πρέπει να ε, δώσουμε μεγαλύτερη ευθύνη και μεγαλύτερη συμμετοχή στον αλληλευτικό κλάδο, σύμφωνα με τον Ολλανδικό μοντέλο. Και χαίρομαι που περιλαμβάνεται πλέον αυτό στην πρόταση. Μόνο έτσι θα εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα του κλάδου. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό τώρα. Ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολιτική για την αλία απαιτεί μακροπρόθεσμους στόχους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαίρομαι που ξεκινάει με την πράσινη βιβλίο, είναι αξιοσημείωτο. Δεν είμαστε κατά, αντίθετα. Δεν θέλουμε να αποτύχουμε πάλι. Δεν θέλουμε μια λάθος πολιτική. Μέχρι τώρα αποτύχαμε γιατί η εφαρμογή της πολιτικής ήταν κακή, όχι γιατί η ίδια η πολιτική ήταν ε, κακή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί η πολιτική πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να τεθεί και σε εφαρμογή, να είναι απλή δηλαδή. Οπότε χαίρομαι με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειοποίηση, περισσότερη συμμετοχή του τομέα και πάνω απ' όλα κανόνες οι οποίοι να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Άκουσα και τον Πορτογάλο συνάδελφο τι είπε για τις διαφορές ανάμεσα στην αλεία και τον ελευθερικό στόχο. Ε, ε, ε, στόλο. Υπάρχει διαφορά βέβαια, μεγάλη ανάμεσα στα δύο. Ο τομέας, οι δύο αυτοί τομείς είναι ξεχωριστοί. Μάλιστα το Σάββατο που μας πέρασε μίλησα με εκπροσώπους του τομείς και επιστήμονες και αλείς συμφωνούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Η γνώση είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε τη σωστή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την εξαίρετη εκθεσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά. Ο κύριος Τσουκαλάστορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ την Επίτροπο κυρία Δαμανάκη και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη συνάδελφη κυρία Μαρία Πατράου Νέβες για την εξαντλητική και εξαιρετική της εργασία. Όλα τα σημαντικά έχουν ήδη λεχθεί. Σε τρία σημεία θα εστιάσω την προσοχή μου. Ένα, σχετικά με την υπεραλίευση. Η υπεραλίευση αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονό. Πράγματι, όπως είπε ο κύριος Αρσένης, εκτιμάται σήμερα ότι έως και το 88% των πληθυσμών στις ευρωπαϊκές θάλασσες απειλούνται από την υπεραλίευση, δηλαδή ελιεύονται σε βαθμό που δεν επιτρέπει την ανανέωσή τους. Η διαχρονική υπεραλίευση έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή αλληλεία σε ολοένα και μικρότερες αποδόσεις, με ταυτόχρονη απώλεια θέσεων εργασίας. Τα ψάρια που αλλιεύονται είναι όλο και μικρότερα, πολλά πριν φτάσουν καν σε αναπαραγωγική ηλικία, ενώ είναι όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Η Ευρώπη αλλιεύει πολύ λιγότερα ψάρια σήμερα από ό,τι πριν από 15 χρόνια, περίπου 25% λιγότερα, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η προσπάθεια και το κόστος αλλιείας. Όμως, κατά τη λήψη μέτρων δεν θα πρέπει να προβούμε σε υπερβολικές αντιδράσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσμενή αποτελέσματα, καθώς όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, σαφώς και έχουμε υπεραλίευση, δεν μιλάμε όμως για κατάρρευση των αποθεμάτων. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι η βιωσιμότητα έχει τρεις διαστάσεις που τονίζει και η έκθεση Νέβες, την κοινωνική, την οικονομική και την οικολογική. Μια αλλιευτική πολιτική που να στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη δεν πρέπει μόνο να ασχολείται με τα ψάρια, αλλά πρέπει να έχει στο επίκεντρό της και τον άνθρωπο. Τα ψάρια, ο άνθρωπος, οι κορμοράνοι και οι φώκες αποτελούν ανταγωνιστικά συστήματα του ίδιου όμως οικολογικού περιβάλλοντος. Τέλος, θα πρέπει να τονίσω την αιμονή μου, όπως και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι είπαν, για την ενίσχυση της αλλιευτικής έρευνας. Και δεν είναι δική μου αιμονή, είναι ε, μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια όσων είπε και ο συνάδελφος κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό τώρα. Η κυρία Τράτμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ όλους τους συζητητές πρώτα απ' όλα για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας και για την τεράστια δουλειά που κάνανε παρόλο που τα συμφέροντα ήταν μερικές φορές αποκλίνοντα. Το Κοινοβούλιο πια μπορεί να μιλήσει περί μιας ε, κατευθυντήρια γραμμής ενός προσανατολισμού που θέλει να έχει η αλία μας στο μέλλον. Έπειτα, κατά τις επραγματεύσεις, προτεραιότητά μας ήταν το κείμενο να ανταποκρίνεται στις ε, ανησυχίες των αλλιέων. Τα καταφέραμε και οι διατάξεις σχετικές με τις ατομικές ε, ποσοστώσεις που μεταφέρονται έχει απαλληφθεί. Τρίτο αποτέλεσμα που θέλαμε ήταν για το μελλοντικό κείμενο να μιλάει για τη συμμετοχή bottom up, από κάτω προς τα πάνω, διαβούλευση με όλους τους φορείς. Επίσης πρέπει να συμπεριλαμβάνει και βασικά στοιχεία όσον αφορά τους σοσιαλιστές όπως είναι η ανθρώπινη και η κοινωνική διάσταση για ολόκληρο τον τομέα συνδυάζοντας αυτά με μια πρακτική βιώσιμη αλίας και διατήρησης των αποθεμάτων. Θέλω επίσης να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Αν θέλουμε να πετύχουμε μια τόσο φιλόδοξη μεταρρύθμιση, πρέπει να αφιερώσουμε στην πολιτική αυτή κονδύλια τα οποία να είναι στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Αυτό θέλουμε μέσα δηλαδή και κονδύλια κατάλληλα για να φέρουμε σε πέρα στην πολιτική μας αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Τραντμένου. διακόπτη ο πρόεδρος, τώρα η κυρία Μπιλμπάου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Δαμανάκη, έχουμε σαφείς στόχους. Θάρρος και δεν θέλουμε να έχουμε ξανά αποτυχία. Πώς? Με τη συμμετοχή. Ο τομέας, η μεταπητική βιομηχανία θέλουν μια βιώσιμη αλία. Γι' αυτό και πρέπει να συμμετέχουν στην σκιαγράφηση της πολιτικής αυτής. Όπως το 2009 που έπρεπε να είχε ετοιμαστεί πιο ανοιχτά. Είναι βασική συμμετοχή λοιπόν για να πετύχει μεταρρύθμιση. Θέλουμε ένα βιώσιμο τομέα, αποδοτικό. Τα υπόλοιπα που είναι σημαντικά είναι η περιφερειοποίηση, η υπευθυνότητα, η σταθερότητα και η δικαιοσύνη. Περιφερειοποίηση διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διατερότητες της κάθε ζώνης. Και είναι άλλο η μικρή κλίμακα και άλλο η βιομηχανική. Έπειτα, θέλουμε καλές πρακτικές. Σταθερότητα με διαχείριση που να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Και τέλος δικαιοσύνη. Να μεταρρυθμιστεί η αγορά και να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται και στις τρίτες χώρες. Δικαιοσύνη επίση για τι γυναίκε που δουλεύουν στη θάλασσα, που είναι αυτέ που συνέχεια ξεχνάμε. Χωρί τη δικιά του τη δουλειά, η αλία σε πολλέ περιοχέ του κόσμου δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Ένα λεπτό τώρα, ο κύριο Βλάσακ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, η πράσινη βίβλος για τη μεταρρύθμιση της κοινή ελληνικής πολιτικής είναι ευπρόσδεκτη. Θέλουμε όντω να απλοποιήσουμε την νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να είναι και πιο αποτελεσματική η νομοθεσία μας. Χαιρόμαστε πολύ για την προσέγγιση της Επιτρόπου να έχει μια πολυετή στρατηγική προκειμένου να διατηρηθούν τα λεφτικά αποθέματα. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί ένα συμβιβασμό ανάμεσα στην Ελία και το περιβάλλον. Η πράσινη βίβλο αποτελεί το πρώτο βήμα σε αυτό το τομέα εν ώψη της μεταρρύθμισης. Αυτό όμως που θα ήθελα να δω είναι να τονίζουμε περισσότερο την υδατοκαλλιέργεια. Να προωθήσουμε λοιπόν και αυτού του είδους ε, την αλία και όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στα εσωτερικά ύδατα και στις παράκτιες περιοχές και να έχουμε καλή ποιότητα τρόφιμα. Ιστηρίζω όλες τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο κύριος Βαλέντσα τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. και Η Αλία, κυρίες και κύριοι, έχει τεράστια σημασία για τις παράκτιες περιοχές και επειδή αποτελεί και πηγή διατροφής για τον κόσμο. Όμω φοβάμαι ότι δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στου στόχου μα. Παραμένουν πολλά προβλήματα. Η υπερβολική εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων, για παράδειγμα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε μια καλή αλλιευτική πολιτική. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Πρέπει όμως να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί. Πρέπει να έχουμε μια πραγματικά αποτελεσματική ε, πολιτική για την αλία. Ε, ευχαριστούμε την εισηγήτρια, κύριε Πατρονένης, για τη δουλειά που έκανε και τα σχόλιά μου είναι τα εξή. Πρώτα απ' όλα, να σταματήσει η υπερβολική εκμετάλλευση των πόρων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα βασικό που πρέπει να λυθεί μέσω μηχανισμών αγοράς, των κατάλληλων μηχανισμών και των ελέγχων βέβαια. Έπειτα, όσον αφορά τα ατομικά συστήματα ποσοστώσεων, επ' αυτού, είναι ένα οικονομικό μέτρο, ένα φάρμακο, ώστε να προσαρμοστεί ο στόλος. Δεύτερον, αποκέντρωση. Είναι πολύ σημαντική επίσης και πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρέπει να φροντίσουμε να αναλάβουν τις υποχρώσεις τους οι αλλοίς από αυτού και να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους αλλοίς. Η πράσινη αυτή βίβλος έρχεται μια πολύ σωστή στιγμή. Γι' αυτό και χρειάζονται και σωστές προτάσεις. Η πολιτική αλλίας δεν είναι τέλεια. Η κυρία Νέβες προτείνει διατάξεις και δυνατότητες για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των αλλιών. Όμω, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται παρετέρω συζήτηση και άλλε προτάσει. Αλλιώ, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει, θα ψηφίσει μια κοινή ελληνική πολιτική που δεν θα λύσει τα προβλήματα τη αλλία στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Ένα λεπτό τώρα. Η κυρία Ιωτόβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που διαμορφώνουμε μια πολιτική μετά την υιοθέτηση της συνθήκης της Αβώνας ε, έχουμε μεγάλες ευθύνες, το αναγνωρίζω. Η συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο ήταν ζωηρότατη και ευχαριστώ την εισηγήτρια γιατί η δουλειά που έκανε είναι πάρα πολύ καλή. Να τονίσω κάποια από τα στοιχεία της μεταρρυθμίσεως που είναι πολύ σημαντικό για όλο τον τομέα. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή της καταστάσεως μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκή Ενώσεως το 2004 και το 2007 και να συμπεριλαμβάνει τα νέα κράτη-μέλη. Το εφιστάμενο σύστημα αναλύσεως και λήψεως αποφάσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη τις νέες υδάτινες επιφάνειες και τις ιδιαιτερότητες θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη που υπάρχει να τονιστεί ο εύξηνο πόντο, η μαύρη θάλασσα, ε, και ειδικό φορέα που θα πρέπει να δημιουργηθεί για τη το διαχείριση του ευξήνου πόντου και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, ο πληθυσμό των παρευξηνίων περιοχών. Και αυτό στα πλαίσια του μελλοντικού οικονομικού πλαισίου που πρέπει να ενταχθεί η μεταρρύθμιση αυτή. Και τέλος, δεν νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση για την μείωση του δυναμικού του στόλου, του πλεονασμού δυναμικού του στόλου, που μπορεί να έχει αρνητικέ συνέπειε όσον αφορά του αλληλεί τώρα την περίοδο τη μεγάλη οικονομική κρίση. Ένα λεπτό, Κρι Ντέιβι. Χωρί μικρόφωνο, μιλητή. Το... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω η Επίτροπο να ενθαρρυνθεί από την ψηφοφορία που έγινε αυτό το μήνα για τον Ιθροτόνο. Θα καταλάβατε τι συναισθήματα επικρατούν στο σώμα και κάποιε ενδείξει ότι μπορείτε να βασιστείτε σε πολλά μέλη εδώ που θα υπερψηφίσουν για ριζικέ μεταρρυθμίσει. Χθε αρκετά μέλη παρέστησαν σε ένα σεμινάριο που διοργάνωσα, μια παρουσίαση από το Συμβούλιο για τη ε, διαχείριση των θαλασσών, το Stewardship Council, δημιουργήθηκε εδώ και 10 χρόνια από σύμπραξη μεταξύ περιβαλλοντολόγων και επιχειρήσεων. Και πάντα είναι καλή αυτή η συνεργασία. Ξεκίνησε αργά, αλλά στο τέλος του έτου, περίπου 10% των αλλιευμάτων θα τύχουν πιστοποίηση από αυτό το φορέα. Αυτό δίνει αξιοπιστία στους πολιτές που υποστηρίζουν το MSC, e, δίνει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και όχι μόνο βάζει περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ψαράδων που έχουν επιστοποίηση για τη βιωσιμότητα των λευμάτων του, δίνει και υπερηφάνεια. Έχουν ένα χαρτί. μπορεί να το δείξουν στι οικογένειέ του και στι κοινότητέ του ότι η σκληρή του δουλειά σημερινή δεν είναι επιβλαβή για τι προοπτικέ τι μελλοντικέ όσον αφορά τα λευτικά αποθέματα. Αυτό συμπληρώνει οδήποτε, η αδίποτε προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ελπίζω η Επίτροπο να υποστηρίξει τι εργασίε του Συμβουλίου. Δημιουργεί πολύ καλά πρότυπα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό τώρα. Η κυρία Μαγκίνε έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια γιατί έκανε πάλι πολύ καλή προσπάθεια, πολύ λεπτομερή προσπάθεια σε αυτό το θέμα. Από την θέση σε ισχύ τη Λισαβόνα, αφού πέρασε η θέση τη Λισαβόνα, θα γίνουν πολύ σημαντικέ μεταρρυθμίσει στον τομέα τη Γεωργία και τη Αλία. Και τα, είναι παρόμοια τα θέματα. Θέλουμε ό,τι καλύτερο για το κάθε τομέα και θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε του τομεί με έναν τρόπο που να δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ανησυχώ κάπως και η συγγήτρια το αναφέρει επίσης στην επισηματική της σημείωση ότι το 2002 εκεί είχαμε καλές προθέσεις αλλά αυτή η μεταρρύθμιση απέτυχε όσον αφορά το ελευτικό τομέα και απέτυχε όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητας. Αλλά βέβαια ενθαρρύνω με τα μάλα από την πολύ πρακτική προσέγγιση που ακολουθείτε τώρα στην προσέγγιση και στις προτάσεις που κάνει, τις τρεις αρχές, περιβάλλον, κοινωνία, ε, και η οικονομία και οι πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και αφορά το τοπικό επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο, ξέρω ποιοι επηρεάζονται, θα ήθελα να πω ότι μου αρέσει το να ψαρεύουμε λιγότερο και όχι περισσότερο και αν το πετύχουμε αυτό μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο και τη γεωργία. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό τώρα, ο κύριος Κάπουλα Ευχαριστώ πρόεδρε. Το έχουν πει πολλοί ομιλητές μέχρι τώρα ότι μια αλία οικονομικά βιώσιμη, αξιοπρεπής κοινωνικά πρέπει να πετύχει. Αυτή πρέπει να είναι η στόχη μας. Η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μια καλή διάγνωση για το ποια είναι τα προβλήματα. Θέτει πολλά ερωτήματα. Διστάζει όμως όσον αφορά τις λύσεις. Η έκθεση επίσης αναφέρεται σε διάφορες ε, αρχές συνενετικές που πρέπει όμως να ερμηνευτούν σε μέτρα στην πράξη και να μπορούν να τηρηθούν. Αυτό πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρέπει επίσης να προσθέσουμε εδώ και τις προσπάθειες που γίνονται στην πρόταση προκειμένου να μπορούν να υπάρξουν και τροποποίησεις στη συνέχεια εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα ή είναι επίμαχα. Η Επιτροπή λοιπόν τώρα στην νομοθετική της πρόταση πρέπει να μας προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να μας επιτρέψουν και μας να θέσουμε σε εφαρμογή τα μέτρα τα οποία εγκρίνουμε χωρίς καμιά αμφιβολία με μεγάλη πλειοψηφία. Σάντσες Πρεσέδο τώρα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής ε, πολιτικής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί από αυτήν εξαρτάται η ζωή πολλών ανθρώπων που ζουν κοντά στις ακτές μας. Επίσης είναι πολύ σημαντική για την ε, ασφάλεια για την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν οι καταναλωτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πολύ σημαντική και για την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη, αηφόρο και ανταγωνιστική αλεία με κοινωνική διάσταση που να σέβεται το οικοσύστημα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την διατήρηση των πόρων και να αναθεωρήσουμε την αρχή της σχετικής σταθερότητας. Το θέμα των ποσοστώσεων τώρα επίσης πρέπει να συμπεριληφθεί. Να αυξηθούν όμως οι έλεγχοι. Ο θέμετος ανταγωνισμός να πάψει να εμφανίζεται στα μέρη μας. Χρειάζεται λοιπόν διαφοροποιημένη μεταχείριση στον τομέα της αλίας και να συμπεριλάβουμε και αυτούς που ασχολούνται με την αλία των κοχυλιών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, των στράχων κλπ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την Επιτροπή και ζητάω και από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε. Τελευταίο στον κατάλογο είναι ο κύριος Κρίστενσεν. Για ένα λεπτό κύριε Κρίστενσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η κοινή η πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά εξίσου σημαντικό είναι η πολιτική αυτή να τύχει της υποστήριξης των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά των εμπλεκομένων φορέων στον κλάδο της ε, αλληλείας. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που τίθεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή διάσταση για να υπάρχει αποκέντρωση των στόχων. Προτού ωστόσο το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολιτική η οποία θα δίνει κίνητρα τους αλληλείς προκειμένου να μειωθεί, να καταργηθεί η λαθροαλία γιατί φυσικά αυτό υποσκάπτει τις προσπάθειες εκείνων που τηρούν τους κανόνες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στα μικρά σκάφη και θα πρέπει φυσικά τα προϊόντα να διατίθενται σε μια λογική τιμή και να ληφθεί υπόψη και το απόθεμα. Πραγματικά χρειαζόμαστε ε, αυτή την μεταρρύθμιση. Με τον κύριο Κρίστησεν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Τώρα περνάμε στο Catch the Eye του Προέδρου. Εφτά συνάδελφοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να παρέμβουν εδώ, κάτω από αυτή τη διαδικασία, ενώ προβλέπονται πέντε. Τώρα πέντε με 7 νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα να δώσουμε το λόγο και στους 7. Αλλά σίγουρα θα σας διακόψω μετά από ένα λεπτό, γιατί ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας μόνο. Η κυρία Σάντσε Σμίθ έχει πρώτα απ' όλα το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να χαιρετήσω εδώ τις ε, προτάσεις της εισηγήτριας για την πράσινη βίβλο. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η νέα στρατηγική πρέπει να προωθήσει μια αλία εγκύτητας. Η δατοκαλλιέργεια αποτελεί μέρος όμως της αλίας από την οποία έχουμε πολλούς πόρους και πολλές θέσεις απασχόλησης. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λοιπόν και ποιοτική υδατοκαλλιέργεια. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας επίσης στην καλλιέργεια οστράκων, κοχυλιών που χρειάζονται και επίσης μια πολύ καλή ανταπόκριση από τη δικιά μας την πλευρά. Η κρίση πλήττει και αυτούς τους τομείς. Οι αλλαγές στο περιβάλλον κάνουν πιο ευάλωτη την παραγωγή μας, περισσότερο ασταθή. Όμως ο κόσμος περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σταθερότητα. Πρώτα απ' όλα μια οικονομική ενίσχυση που να τους επιτρέπει να ζήσουν από την παραγωγή τους και έπειτα ε, μεταβατική ενίσχυση ώστε να μπορέσουν οι πόροι αυτοί διακόπτει ο πρόεδρος ο κύριος Άλβες τώρα έχει το λόγο έλεξε ο χρόνος σας Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα παρακαλώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους αλείς από τις αζόρες που έχουμε εδώ στα θεωρία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που συμπεριέλαβε στην έκθεσή της και ειδικά μέτρα για τις άκρος περιφερειακές περιοχές. Ζητάει να ληφθεί υπόψη επίσης η παράκτη αλία. Θέλω Επίσης να υπενθυμίσω και τις τροπολογίες της σοσιαλιστικής ομάδας που εγκρίθηκαν από την εισηγήτρια και που οι διάφορες ενώσεις αλλιέων από τις Αζόρες θέλουν να υιοθετηθούν. Εμείς από τις άκρως περιφερειακές περιοχές θέλουμε βιογραφικές περιοχές ώστε να προωθήσουμε τους υπάρχοντες πόρους. Και είναι αναγκαίο αυτό εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τις θαλάσσιες περιοχές Οπότε πρέπει να ξαναδούμε και να θεωρήσουμε το όριο των 6 μιλίων 18. κόβει ο πρόεδρος. Κύριος Λέιον, το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω να, συγχαρώ να συγχαρώ την εισηγητρία. Η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία έχει υποστεί πλήγματα και αυτή η μεταρρύθμιση μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια νέα αρχή. Μου φαίνεται ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να κερδίσει το γόητρο που της αξίζει, θα πρέπει όμως να έχει τη βιωσιμότητα που, που, τη, που χρειάζεται. Κατά δεύτερον, τη σταθερότητα που χρειάζεται και προβλεψιμότητα σε ό,τι αφορά όλο τον κλάδο. Έτσι, αντιμετωπίζοντας την υπεραλίευση, θα πρέπει να βρεθεί μία λύση για την υπερβολική αυτή παραγωγή. Θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειες του παρελθόντος και θα πρέπει να βρούμε μία πραγματική λύση στο θέμα των απορρίψεων. Επί της ουσίας, η μεταρρύθμιση της κοινής αλευτικής πολιτικής θα πρέπει να δώσει ένα μέλλον στον αλευτικό κλάδο και στους αλληλείς. Επί της ουσίας θεωρώ ότι το κλειδί και διακόπτει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ρωμέβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να αποφελθώ από την ευκαιρία αυτή για να επιμείνω στα σημεία εκείνα που πολλοί από εμά πιστεύουν ότι είναι ζωτική σημασία για την έκθεση που θα ψηφίσουμε. Υπενθυμίζω λοιπόν ποια είναι αυτά τα σημεία. Πρώτα απ' όλα, η πρόληψη είναι κάτι πολύ βασικό. Η αρχή τη προφύλαξη δηλαδή. Έπειτα, όχι υπερβολική ελίευση. Ε, Περιορισμό ε, των ε, δημοσίων ενισχύσεων. Βελτίωση του ελέγχου και δίωξη των παραβάσεων. Χωρί εξαιρέσει γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνέπειες και κυρώσει για αυτόν που κάνει αυτό που δεν πρέπει. Συγχρόνω όμως να ενισχύσουμε την βιώσιμη αλεία. Να προχωρήσουμε στον ορισμό. Τι είναι μικρή κλίμακα αλεία. Είναι πολύ βασικό και αυτό. Χρειάζεται διευκρίνηση. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ και να ζητήσουμε περισσότερη συνοχή στις συμφωνίε της αλλιευτικέ με τρίτες χώρες. Μαρόκο και για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Κούν έχει τώρα το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο, κυρία Δαμανάκη και τη εύχομαι καλή τύχη και θα ήθελα να πω προ την κυρία Νέβε ότι είναι εξαιρετική η εργασία τη και είναι σημαντικό να αποτυπώνονται και οι ανάγκε των μικρών ε, αλλιευτικών κρατών και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για τη Γερμανία. Φυσικά όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι τα ήχθη από θέματα θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και να τα καταστήσουμε βιώσιμα αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον για του αλλιεί μα. Αλλά όχι μόνο να λέμε ότι συζητάμε συζητάμε οικονομικά και οικολογικά θέματα. Όχι, να συζητήσουμε για ε, απειλούμενα είδη, να δούμε τι γίνεται με τις κορμοράνους για παράδειγμα. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμή και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ότι εκπροσωπεί αυτή, αυτό, αυτή η ακτογραμμή οικογένειες που εξαρτώνται για τη διαβίωσή τους ε, από την άλλη Είναι καλή λοιπόν αυτή η πράσινη βίβλος και διακόπτει εδώ η πρόεδρος. Η κοινή ελευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και οικονομικά θέματα αλλά και περιβαλλοντικά θέματα και όλα αυτά να τα εναρμονίζει με τις ανάγκες διαβίωσης των αλλιέων. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν τα αποθέματα και να διαμορφωθούν βάσει των επιστημονικών κριτηρίων. Χρειαζόμαστε λοιπόν υποστήριξη του ελευτικού κλάδου και μάλιστα από πολλές απόψεις στις επενδύσεις, στον συγχρονισμό, στην ε, κοινωνική διάσταση. Η κοινή ελευτική πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, τις συγκεκριμένες ε, συνθήκες που επικρατούν σε κράτη-μέλη, σε περιφέρειες αλλά και θάλασσες. Και φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θέματα συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και των τοπικών αρχών. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη συμμετοχή και στους ίδιους τους αλληλείς και να τονωθεί η αλυσίδα από τον αλληλέα μέχρι τον καταναλωτή. Ο το Κατά τη διάρκεια των 7 μηνών θητείας σαν Ευρωβουλευτή, ποτέ δεν συνάντησα επιθυμωμένους ανθρώπου από τους αλληλείς και τις γυναίκες αλληλείς που συνάντησα στην ε, εκλογική μου περιφέρεια. Η κοινή αλληλευτική πολιτική δεν λειτουργήσε για αυτούς οπότε μεταρρύθμιση είναι άκρο ευπρόσδεκτη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τα λευτικά αποθέματα, πρέπει να διατηρήσουμε και τι παράκτιε κοινότητε και τα δύο δεν αποκλείουν το ένα το άλλο απαραίτητα. Χρειάζεται να υποστηρίξουμε του μικρού ε, αλληλεί. Και όπω αναφέρθηκε από τον κύριο Μπόντ, νέα τεχνολογία θα πρέπει επίση να χρησιμοποιηθεί, κυρίω αυτά που αναφέρθηκαν, για να κάνουμε μεγάλη διαφορά και το θέμα της έρευνας θα πρέπει να εξεταστεί. Όταν ακούμε έρευνα, Θεωρούμε να εμπιστευόμαστε και τα επιστημονικά στοιχεία χωρίς να τα αφισβητούμε. Θα πρέπει λοιπόν όμως αυτά να είναι πολύ επίκαιρα στοιχεία και να είναι ενήμερα. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνέδαρφε. Τελειώσαμε τον κατάλογο ομιλητών για τον κύκλο αυτό παρεμβάσεων. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαρτίν Φραγέιρο, ο οποίος εκ μέρους του Συμβουλίου θα αντιδράσει στις διάφορες παρεμβάσεις που ακούστηκαν εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Μαρτίν Φραγέιρο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πατράο Νέβες, την εισηγήτρια, για τη δουλειά της. Μέχρι τώρα στις συζητήσεις στο Συμβούλιο πρέπει να σας πω ότι οι Υπουργοί στηρίζουν ομόφωνα την μεταρρύθμιση, θέλουν απλοποίηση, συνοχή στους κανόνες και ενίσχυση των ελέγχων σε περιφερειακό επίπεδο Λαμβάνοντα υπόψη όλα τα στρατηγικά στοιχεία. Συμφωνούν για το ότι πρέπει να μειωθούν ε, τα ψάρια που επιστρέφουν στη θάλασσα, που τα πετάμε, τις απορρίψεις. Όσον αφορά τα 12 μίλια, είναι κάτι που συζητάμε. Το θέμα της συμμετοχής επίσης των, ε, όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στον τομέα αυτό ενίσχυση των εσόδων των αλλιών, συζητάμε επίση επιδοτήσεις ως μέτρο όμω έκτακτα. Ναι, για την έρευνα, για την υδατοκαλλιέργεια, για την σχέση της κοινή ελευτική πολιτικής με την ολοκληρωμένη μας πολιτική για τη θάλασσα και για τις ελευτικέ συμφωνίες. Μέχρι τώρα οι συζητήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι υπάρχουν αποκλήσεις όσον αφορά ορισμένες πτυχές το θέμα των ποσοστώσεων, της μεταβίβασης των ποσοστώσεων, ο περιορισμός της προσπάθειας, η μέθοδος για να μειώσουμε τις απορρίψεις, η υπεραλίευση, η χρηματοδότηση, όπως επίσης και η αύξηση της ενίσχυσης για την αλία μικρής κλίμακας και παράκτειας. Το Συμβούλιο μέχρι τώρα δεν έχει καταλήξει σε θέση. Δεν προβλέπεται να υιοθετήσει κάποια απόφαση πριν από την επόμενη χρονιά, περιμένει πρώτα την επίσημη παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να χαιρετήσω και εγώ εδώ τους αλείς, τους εκπροσώπους των αλλιών που βρίσκονται εδώ στα θεωρία. Ευχαριστούμε κύριε Μαρτίν Φρεγέρο. Η κυρία Δαμανάκη έχει τώρα το λόγο. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για την ε, συνεισφορά τους είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι έγιναν τόσες πολλές παρεμβάσεις. Η βιωσιμότητα αναφέρθηκε εκτενώς. Οπότε συμφωνούμε ότι είναι ένα πλαίσιο γενική συμφωνία η βιωσιμότητα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα όσα εθίγησαν. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποιες προτεραιότητες. Αλία μικρής κλίμακας και παράκτιες περιοχές αποτελούν προτεραιότητα. Σας διαβεβαιώνω όλους σας ότι θα πάρουμε πολύ στα σοβαρά αυτά που μας είπατε σχετικά με το θέμα. Επίσης, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω πρόθεση να λάβω σκληρά μέτρα για τους ερασιτέχνες ψαράδες μετά, περιφερειοποίηση, δεύτερη προτεραιότητα. Θα ήθελα πολύ να συζητήσω λεπτομερέστερα τι ακριβώς κάνουμε για να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή. Διότι εδώ γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα. Μεταφερόμενα ληφτικά, μεταβιβαζόμενα ληφτικά δικαιώματα. Από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ ε, αγαπημένο θέμα συζητήσεων αυτό, με πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στη ψηφοφορία. Θα ήθελα να πω όμως ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πρόβλημα αυτό. Πολλά κράτη-μέλη εφαρμόζουν το σύστημα ήδη. Τι προτείνω λοιπόν. Να διεξαχθεί μια συζήτηση ίσως και στα πλαίσια της Επιτροπής Αλίας. Εφόσον δεν λύγει εδώ διάλογος, μπορεί να διεξαχθεί μια συζήτηση για τα μεταβιαζόμενα δικαιώματα, τα ληφτικά δικαιώματα. Βλέπω και την κυρία Φράγα που είναι εδώ, μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε το θέμα. Κάποιες άλλες προτεραιότητε, να αναφέρω τώρα. Ισότιμες συνθήκε για την περιοχή τη Μεσογείου και του αλληλεί άλλων χωρών ε, σωστό πρέπει να το κάνουμε αυτό, να υπάρξει συμφωνία μαζί τους για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των δικών μας αλλιέων και εκείνων. Η εξάλληψη των απορρίψεων, η σήμανση προτεραιότητες και αυτές. Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη για νέα μορφή αλλιευτικών συμφωνιών. Νέα μορφή που θα συμπεριλαμβάνει τη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας στη συζήτηση και πιστεύω ότι δεν λύγει εδώ ο διάλογος. Ξεκινά μια άριστη συζήτηση μεταξύ μας εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τελειώνουμε με το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης, δίνοντας το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Πατράου Νέβες, για δύο λεπτά. Έχει ένα ωραίο όνομα. Πατράο Νέβε. Ναι, συνδυάζει τη γη με τον ουρανό. Μαρία Ντεθέο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους όσοι σήμερα έλαβαν το λόγο στην ε, Ολομέλεια και που παρουσίασαν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την διαδικασία αυτή γιατί όπως είπε και η κυρία Επίτροπο, θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει σε αυτή τη μακρά διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι με μία έκθεση δεν μπορούν να συμφωνήσουν ασφαλώς όλοι, αλλά καταφέραμε να πετύχουμε αρκετά. Ίσως κάποιοι βέβαια να κρίνουν ότι δεν προχωρήσαμε ως προς την επίτευξη των στόχων μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με την έκθεση αυτή καταφέραμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των βασικών ερωτηματικών και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και μια συνένεση για να απαντήσουμε στις απαιτήσει οι οποίες ε, τίθενται από τον ε, αλλιευτικό κλάδο στην, στην Επιτροπή Αλληλείας εργαστήκαμε υπό την Προεδρία της κυρίας Φράγκας και ελπίζω να συνεχιστούν οι εργασίες ε, στα πλαίσια της Επιτροπής μας και να μπορέσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεργαστούμε, να συνεχίσουμε αυτή την συνεργασία προκειμένου να επεξεργαστούμε και τις νομοθετικές προτάσεις. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας, θα καλυφθούν με ισορροπημένο τρόπο όλα τα θέματα για την μεγάλη και πολυδιάστατη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα βρούμε απαντήσεις για τα θέματα που πλήττουν την ε, αλευτικό κλάδο. Αν το καταφέρουμε λοιπόν αυτό, θα έχουμε επιτελέσει και ένα μεγάλο έργο υπέρ του αλευτικού κλάδου. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να εγγυηθούμε την βιωσιμότητα του κλάδου σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Ευχαριστούμε την εισηγητρία. Κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει σε μία ώρα, στις 11.30. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης, που είναι η δήλωση της Επιτροπής για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Σήμανσης είναι ένα σημείο το οποίο βέβαια είναι πολύ επίκαιρο δυστυχώς γιατί ακριβώς εδώ στις